για τα νέα έργα, τι νέε δραστηριότητε που θα ξεκινήσουμε στις στα πλαίσια τη στρατηγική του Δούναβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση που αφορά το διαμεσολαβητή. Η κυρία Ματσόνη έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πως κάθε χρόνο και φέτος προσπαθούμε να προβούμε σε έναν απολογισμό της δραστηριότητας του διαμεσολαβήτη. Υπενθυμίζω ότι ο διαμεσολαβητής δυνάμει του άρθρου 298 μπορεί να δράσει και μέσα στα πλαίσια του δικτύου διαμεσολαβητών έτσι ώστε να τηρούνται, ε, μάλλον να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών δυνάμει του άρθρου 46 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δηλαδή, ο καθένας θα μπορεί και, θα, μπορεί και πρέπει να την χάνει ίσης μεταχείρισης εξ ονόματος ε, εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται τάχιστα. Σήμερα Είχαμε περισσότερες φέτος από 2.100 είχαμε περίπου 2.600 καταγγελίες και το νέο στοιχείο είναι ότι το, 16, το 61% χρησιμοποίησε το ίντερνετ και μέσα στα πλαίσια αυτού το 61% το 53% έγινε με βάση μία φόρμα που ε, υποβάλλεται, που υπάρχει στον ιστότοπο. Και η Επιτροπή Αναφορών θα ήθελε να υπάρχει μία υπηρεσία διαδικτύου έτσι ώστε και η δική μας σελίδα να είναι πιο προσιτή στον πολίτη το 2011 μειώθηκαν ε, οι, τα αιτήματα πληροφόρησης γιατί ο οδηγός του διαμεσολαβητή ήταν σαφός και έτσι μειώθηκαν οι αιτήσει πληροφόρησης ή διασαφήνισης. Επίσης μειώθηκαν και τα σφάλματα παρουσίασης γιατί πολλές φορές τα αιτήματα δεν είχαν διατυπωθεί σωστά ώστε να εμπίπτουν στο, στην εντολή του διαμεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής προσπάθησε να διευκολύνει τους πολίτες και ως προς τη διαδικασία του 11 είχαμε και ένα πλαίσιο απλούστευσης. Βεβαίως, αυτή η χρηστή πρακτική βοήθησε στο να υπάρχει καλύτερη παρουσίαση και οι υπηρεσίες να είναι καλύτερες από πλευράς διαμεσολαβητή. Ο αριθμός καταγγελιών όμως παραμένει υψηλός είναι και το υψηλότερο ποσοστό, το 58% δηλαδή. Βεβαίως μπορεί να υποθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια του εκτελεστικού της χαρακτήρα αποτελεί στόχο των πολιτών, αλλά αυτό δεν ε, αποδεικνύει δεν στοιχειοθετεί το βασικό στοιχείο, όπως θα μας πει και ο κύριος Σεύκοβιτς. Έχουν μειωθεί οι καταγγελίες έναντι της Επιτροπής, ενώ αυξάνονται έναντι του Συμβουλίου. Είχαμε 382 καταγγελίες, από αυτές έχουν διαλευκανθεί οι 318. μέσα στα πλαίσια του δικτύου δικαιωμάτων των πολιτών. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συστάσεις προς το διαμεσολαβική. Τι όμως ανταποκρίθηκε αρκετά καλά στο έργο του σε γενικές γραμμές. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διαμαντούρος έχει το λόγο. Με μεγάλη μας χαρά σας ξαναβλέπουμε ένα χρόνο μετά. Μετά από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και βλέπουμε ότι χαίρουμε άκρα υγεία και εσείς και εγώ μετά από τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και είναι εδώ πέρα και ο Επίτροπος Υγείας. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ στην ετήσια μου έκθεση για το έτο 2011. Πρώτα απ' όλα να πω πως είμαι ευγνώμων για την ε, συνεχιζόμενη στήριξη του Κοινοβουλίου στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επίσης να ευχαριστήσω την, ευχαριστίε μου στην πρόεδρο τη Επιτροπή Αναφορών, την κυρία Ματσόνη, για την ε, έκθεση την οποία μόλις ακούσαμε όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει η στήριξη του Κοινοβουλίου και η συνεργασία της Επιτροπής Αναφορών συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή. Αναφερθώ τώρα στα βασικά στατιστικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του 2011 έλαβα ένα σύνολο 2.510 καταγγελιών από πολίτες, εταιρείες, ΜΚΟ, ενώσεις και λοιπούς καταβάλω κάθε προσπάθεια να βοηθήσω κάθε καταγγέλλοντα που απευθύνεται στον διαμεσολαβητή, ακόμα και σε περιπτώσει που δεν εμπίπτουν εντό τη εντολή μου. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το πόσο σημαντικό είναι για του πολίτε να ε, έχουν κάποιον ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στον κατάλληλο μηχανισμό και φορέα από την αρχή και να μην έχουν τις καθυστερήσεις και απογοήτευση όταν ε, προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο θεσμικό όργανο από μόνο τους. Τον Ιανουάριο του 2009 στην ε, ιστοσελίδα μας ε, ξεκινήσαμε έναν διαδραστικό οδηγό και στις 23 επίσημες γλώσσες. Ο οδηγός αυτός έχει στόχο να κατευθύνει τους ε, καταγγέλλοντες στον, στον κατάλληλο φορέα, είτε είναι οι δικέ μας υπηρεσίες, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, η Εθνική Περιφερειακή διαμεσολαβητές ε, των κρατών μελών ή φυστάμενοι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ε, η σελίδα Georg Europe ή το δίκτυο Solvit. Ο αριθμός ε, των καταγγελιών που δεν έγιναν δεκτές έπεσαν και το 2011. Αυτή τη φορά ήταν 111 τον αριθμό. Αποδεί το γεγονός αυτό στον διαδραστικό μας όδηγο καθώς τώρα πλέον οι πολίτες ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν απευθείας το 2011 πάνω από 18.000 άτομα έλαβαν σύμβουλοι από αυτόν τον οδηγό. Αν μετρήσουμε τον αριθμό των ετοιμάτων για πληροφορίες που απαντήθηκαν μπορούμε να πούμε πως πάνω από 22.000 πολίτες βοηθήθηκαν άμεσα από τον διαμεσολαβητή. Επιπλέον η ιστοσελίδα μας είχε πάνω από 295.000 μοναδικές επισκέψεις σε αντίθεση με τη μείωση των, του αριθμού των ετοιμάτων εκτός της εντολής μας, ο αριθμός των ερευνών που ξεκινήσαμε το 2011 αυξήθηκε στις 396, δηλαδή είχαμε αύξηση κατά 18%. Αυτό επιβεβαιώνει πόσο στρέφονται πλέον στο διαμεσολαβητή το κάνουν για τον κατάλληλο λόγο. Ο μεγάλος αριθμός ε, των ε, ερευνών που ξεκινήσαμε είναι και αποτέλεσμα των διαδικασιών των δικών μας, τις οποίες αλλάξαμε για να γίνουν πιο φιλικές προς τον πολίτη. Έχουμε έναν νέο τύπο έρευνας ε, στις, στον οποίο, με τον οποίο επιτρέπουμε να υπάρξει μια διευκρίνηση της καταγγελίας σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε αρχικά πιστεί πως υπάρχουν λόγοι να ζητήσουμε την γνώμη κάποιου θεσμικού οργάνου. Επίσης, έχουμε περαιτέρω στοιχεία για το ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απαντούν θετικά στη στάση μου και ότι παίζουν πλέον ένα πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση των καταγγελιών. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι βελτιωμένη και προτιμητέα σχέση με το παρελθόν, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια ο αριθμός των επικριτικών παρατηρήσεων ήταν πάν, μόλις πάνω από τους 34, ενώ ο μέσος όρος ε, της περίοδου 2006-2008 ήταν μόλις πάνω από 46. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, και φέτος ε, έχω τονίσει κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις για να τονίσω την υποδειγματική αντιμετώπιση από την διοίκηση και τα θεσμικά όργανα κάποιων περιπτώσεων για να τονίσουμε πως η βασική λειτουργία του διαμεσολαβητή είναι να ενισχύσει μια κουλτούρα υπηρεσίας ε, στα θεσμικά όργανα ενισχύοντας ε, τις βελτιστές πρακτικές. Τέτοιες, ε, δέκα τέτοιες περιπτώσεις τονίζονται στην φετινή έκθεση. Η θέληση των θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν με τον διαμεσολαβητή για να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση των καταγγελιών νομίζω πως δείχνει το πόσο δεσμευμένη είναι σε μια τέτοια κουλτούρα η άνθρωποι στις υπηρεσίες. Επίσης, ε, ορισμένες φορές και οι ίδιοι καταγγέλλονται συνεισέφεραν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αμοιβαίως επωφελές. Σύμφωνα λοιπόν με μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου όσον αφορά την απόδοση της Ευρωπαϊκής ε, Διοίκησης, ε, αυτό το οποίο θεωρούσαν σημαντικότερο ήταν το δικαίωμα να διακινούνται και να κατοικούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το 48% και ήταν το δικαίωμα χρηστής διοίκηση, γύρω στο 33% το οποίο ήταν δεύτερο, μαζί με το δικαίωμα να απευθύνονται στον διαμεσολαβητή, 32%. Από την άλλη, 42% είπαν πώ δεν ήταν ικανοποιημένοι με τη διαφάνεια στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52% είπαν πως ο διαμεσολαβητή πρέπει να φροντίσει οι πολίτε να ξέρουν τα δικαιώματά του και πώ μπορούν να τα ασκήσουν. Το 2011 λοιπόν, ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προτεραιότητες, ε, διοργάνωσε τη μεγαλύτερη εκδήλωση ενδιαφερομένων που έχει οργανώσει ποτέ ο Δήμος Ολαβητής με τίτλο εάν η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αποτελέσματα για τους πολίτες. Οι ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων ο κύριος Χέρμαν Φαναρομπόη, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τότε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Νταϊάννα Γουόλης και η κυρία Βιβιάν Ρίτινγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το 2011 δημοσίευσα ένα φυλάδιο με τίτλο «Προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει». Είναι αυτή η έκδοση, δίνει πληροφορίες για όλο το φάσμα μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων ε, στα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζήτηση για αυτό το φυλάδιο ήταν η υψηλότερη για από οποιαδήποτε άλλη έκδοσή μας. Δεδομένης της ε, δυσαρέσκειας όσον αφορά τον βαθμό διαφάνειας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας για το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει τις 28 Σεπτεμβρίου καλώντας την ε, διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση και να υιοθετήσει αρχεία εγγράφων τα οποία θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Επλέον, όσον αφορά τις υπηρεσίες μου ξεκίνησα να δημοσιεύω στην ιστοσελίδα μου πληροφορίες για νέες έρευνες μόλις ξεκινήσουν. Έτσι γίνεται ευκολότερο να παρακολουθεί κανείς την πρόοδό τους από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2009 υιοθέτησα μια δήλωση για την αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η οποία είναι ω εξή. Ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αναζητά δίκαια αποτελέσματα στι καταγγελίε κατά των ε, θεσμικών οργάνων τη Ένωση, ενθαρρύνει την διαφάνεια και προωθεί μια κουλτούρα τη διοίκηση. Σκοπεύει να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη μέσω του διαλόγου των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προαγάγει τις υψηλότερες προδιαγραφές και ε, την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Για να εφαρμόσουμε λοιπόν αυτή την δήλωση υιοθετήσαμε μια στρατηγική. Τα βασικά σημεία της στρατηγικής είναι πρώτον να ενισχυθεί ο διάλογος με τους καταγγέλλοντες στην κοινωνία των πολιτών κλπ. σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην συνθήκες Λισαβόνας. Δεύτερον, να βρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές από συναδέλφους διαμεσολαβητές ε, μέσω μεταξύ άλλων του δικτύου των διαμεσολαβητών και τρίτον ενίσχυση του ρόλου του διαμεσολαβητή στην προώθηση μιας διοικητικής κουλτούρας στα ε, θεσμικά όργανα. Για να υπάρχει λοιπόν χρηστή διοίκηση, ένα βασικό στοιχείο του να είμαστε φιλικοί προσπολίτες στα θεσμικά όργανα και, και ε, οι φορείς πρέπει να αναπτύξουν μια κουλτούρα εξυπηρέτησης των πολιτών. Ένας φορέας λοιπόν που θα έχει μια τέτοια κουλτούρα θα ενθαρρύνει τους ε, υπαλλήλους του να το κάνουν αυτό όχι μόνο επειδή το απαιτεί ο νόμος αλλά να είναι και ευγενικοί και να βοηθούν τους πολίτες θα εξηγούν την λογική και το σκεπτικό πίσω από τις δραστηριότητες τους και θα δέχονται δημόσια εξέταση της συμπεριφοράς τους. Έχοντας αυτά κατά νου, συμπέρανα πως θα ήταν χρήσιμο να βγάλουμε ένα έντυπο το οποίο θα περιέχει με τρόπο συνοπτικό αυτές τις αρχές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι αρχές της δημόσιας διοίκησης δημοσιεύτηκαν στις 19 Ιουνίου φέτος. Θα ήθελα λοιπόν να τι αναφέρω εν συντομία. Πρώτον, αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πολίτε τη. Δεύτερον, ακαιρεότητα. Τρίτον, αντικειμενικότητα τέταρτον σεβασμός για τους άλλους και πέμπτον διαφάνεια. Και είμαι ευγνώμων στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού για το ότι φρόντισε να διανεμηθούν όλα αυτά σε όλους τους εργαζόμενους του Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, όπως έχω επανειλημμένα πει, η δήλωση αυτή για τις ε, αρχές της δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι ούτε η πρώτη βεβαίως, ούτε η τελευταία λέξη και πρόβλεψη όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές συμπεριφοράς που ισχύουν ε, για την ε, Δημόσια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Εδώ πέρα λοιπόν δεν σκοπεύουμε να έχουμε κάποιες νέες προδιαγραφές, απλά να αποσαφηνίσουμε τις προδιαγραφές και των υπαλλήλων και των πολιτών για να έχουμε μια καθημερινή πραγματικότητα για να γίνουν καθημερινή πραγματικότητα οι αρχές οι οποίες ήδη τηρούνται από την δημόσια διοίκηση της Ένωσης. Η προσθέμενη αξία είναι το να ξεκινήσει μια συζήτηση και να υπάρχει ένα αντικείμενο συζήτηση μεταξύ και των υπαλλήλων και του κοινού για την συμπεριφορά η οποία θα είναι ε, η αρμόζουσα. Οι αρχές αυτές δεν έχουν στόχο να επαναλάβουν μέσα τα οποία ήδη υπάρχουν ούτε να υποκαταστήσουν την ε, αναθεώρηση και συμπλήρωση αυτών των μέσων. Ε, θεωρώ όμως πως θα πρέπει να αποτελέσουν μια πηγή ιδεών έτσι ώστε από κοινού με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα η οποία θα καταστήσει σε αυτές τις αρχές μια ζώσα πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντούρου. Εξ της ε, Επιτροπής έχει το λόγο ο κύριος Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητέ κύριε Διαμεσολαβητή. Πρέπει να πω ότι είναι ευπρόσδεκτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πολύ ολοκληρωμένη έκθεση κυρίας Ματσόνη. Θέλω να την συγχαρώ, όπως και την Επιτροπή Αναφορών, για το πολύ σημαντικό αυτό έργο η έκθεση, δίνει μια, η έκθεση του Διαμεσολαβητή δίνει μια πλήρη και εξαντλητική παρουσίαση του έργου του Διαμεσολαβητή το τελευταίο ε, έτος και επίσης βοηθά και τα άλλα ε, θεσμικά όργανα. Μας θυμίζει ότι πρέπει να είμαστε ένας, ε, μια ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση ε, εις όφελος των πολιτών μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά τον κύριο Διαμαντούρο για την εξαιρετική συνεργασία μας και για τη βοήθεια που προσέφερε στο να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Οι προτάσεις του και οι παρατηρήσεις του είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτες και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υπηρεσίας. Ακούστηκαν πολλά νούμερα, πολλοί αριθμοί από την κυρία Ματσόνη και από τον κύριο Διαμαντούρο και θα ήθελα να τα αναφέρω και εγώ μερικά. Πράγματι, ο, διαμεσο, τα αιτήματα προς τον διαμεσολαβητή κυρίως στρέφονται προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 58% ε, το 2011, λίγο κάτω από ότι το 2010 που ήταν 65%, ε, ήταν λίγο λιγότερο το 65%. Αλλά είναι φυσιολογικό σε μεγάλο βαθμό αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, όπως είπε και η συγγήτρια, το μεγαλύτερο θεσμικό όργανο που έχει εκτελεστικές εξουσίες και άρα είναι απολύτως φυσικό να απευθύνονται κυρίως τα αιτήματα ε, προς αυτήν. Πώς αντιμετωπίσαμε όμως ε, τα παράπονα και τις περιπτώσεις που χειρίστηκε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή έστειλε 365 ε, απαντήσεις το 2011 ε, σε σχέση με 375 το 2010. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, τη σημασία του φιλικού διακανονισμού και προσπαθούμε αν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε, περιστα... σε συνθήκες όπου όλοι είναι κερδισμένοι και πιστεύω ότι συμφωνείτε και εσείς ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε. Επίσης, ο αριθμός των επικριτικών παρατηρήσεων ε, έφτασε μόνο το 11% όλων των ετοιμάτων που έκλεισαν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε 25 απαντήσεις προς τον Ευρωπαϊκό δια... στις ε, επικριτικές παρατηρήσεις του ε, διαμεσολαβητή και εν μέρη η πλήρως συμφωνήσαμε σε 18 περιπτώσεις 72% επιπλέον. Ο αριθμός των άτυπων ε, διαδικασιών του 2011 ήταν 99, δηλαδή ε, σημαντική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ε, διαμεσολαβητής ζητά από την Επιτροπή να απαντήσει απευθείας στους πολίτες χωρίς να αναλύσει το περιεχόμενο της απάντησης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον διαμεσολαβητή που οργάνωσε το σεμινάριο αυτό, αλλά επίσης και την πολύ ευρύ αυτή δημόσια διαβούλευση για τις αρχές της δημόσιας υπηρεσίας προς την οποία συνεισφέραμε ε, μέσω του Προέδρου του κυρίου Μπαρόζο. Θέλω επίσης να επιβεβαιώσω ότι ε, εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που τις θεωρούμε σημαντικές και δίνουμε έμφαση στο ότι παρότι ο κανονισμός του προσωπικού επιβάλλει ε, όλα αυτές τις αρχές στα στελέχη και είναι αφοσιωμένη σε αυτές τις αρχές της διοίκησης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σεβόμαστε τον κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς οι αρχές αυτές θα εφαρμοστούν σε όλη την Επιτροπή θα διανεμηθούν στα στελέχη μας και στην εσωτερική εσωτερική και στην εξωτερική ιστοσελίδα μας. και θέλω να καταλήξω επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην ε, συνέχιση και ενίσχυση της εξαιρετικής συνεργασίας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, την Επιτροπή Αναφορών, με πολύ παραγωγικό τρόπο. Ευχαριστώ. για λεπτά κύριος Γιάρ. <clears throat> Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεμαντούρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την καλή του δουλειά και την καλή συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών. Τα νούμερα τα οποία αναφέρατε είναι σατή 2011-2510 ε, 2.510 ε, ε, καταγγελίες Επίσης για εμένα σημαντικό ήταν ε, ο μικρός αριθμός καταγγελιών οι οποίες ε, δεν έγιναν δεκτές γιατί βεβαίως ε, αγωνιζόμαστε και για μια καλύτερη σχέση με τους πολίτες και συγχαρητήρια και για αυτό το νούμερο. Για μένα λοιπόν τα νούμερα αποδεικνύουν πως ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά ο Δημοσιολαβητής προσφέρει στους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημείο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν αν ε, θεωρούν πως ε, δεν τους συμπεριφέρθηκαν δίκαια ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άρα συνεισφέρει στο να γίνει η Ευρώπη πιο απτή και κατανοητή από τους πολίτες μας. Πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε πως ο διαμεσολαβητής δεν είναι μια υπηρεσία χωρίς δόντια Ε, και εδώ πέρα δεν θέλω βεβαίω να ισχυριστώ πω η Κομισιόν τρέμει ενώπιον του διαμεσολαβητή, αλλά νομίζω πως υπάρχει αμοιβαίως σεβασμός και νομίζω πως είναι αυτός ένας καλός τρόπος εργασίας. Ιδιαίτερα με χαροποιεί το ότι η συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπής Αναφορών και του διαμεσολαβητή είναι, θα έλεγα, ιδανική το δικαίωμα του αναφέρεστε και το δικαίωμα να για κανείς των ε, διαμεσολαβητή νομίζω ε, είναι συμπληρωματικά. Το έχουμε αυτό στην πολιτική και βεβαίως ε, συχνά καμιά φορά υπάρχουν και διαφωνίες όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στην περίπτωσή μας και νομίζω πως θα μπορούσε και το σύνθημα του Δημοσιολαβητή να είναι σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία είμαστε υπέρ του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίως και εύχομαι να συνεχίσετε την καλή σας δουλειά και βεβαίως πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για 1,5 λεπτό κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Διαμεσολαβητή, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο για μία έκθεση η οποία είναι ουσιώδης και αναγνωρίζει τη συνεισφορά του ρόλου του. Χαιρόμαστε για αυτή την υποστήριξη και βλέπουμε ότι η Επιτροπή είναι ένας από τους βασικούς σας στόχους έρευνας αυτό που έχει σημασία είναι η χρηστή διοίκηση, η βελτίωση του πλαισίου χρηστής διοίκησης και αυτό ακριβώς επιδιώξαμε ως Επιτροπή Αναφορών όχι μόνο το 2011 αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του, της θητείας σας. Μιλάμε για ένα 58% των ερευνών που έχει στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το 2012 υπάρχουν περιπτώσεις και υποθέσεις που ε, σχετίζονται με τη μη διαφάνεια του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Διαμεσολαβητά και ελπίζω να πείσετε και τους εθνικούς συνήγορους ότι έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Από τους φιλελεύθερους η κυρία Γιατεμάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ομάδας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο για την πολύ καλή του δουλειά στον τομέα της ε, διαφάνειας και για το ότι φροντίζει να υπάρχει ορθή διοικητική πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, εκδώσατε έναν ε, οδηγό σχετικά, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Ε, εξάλλου αυτό τον οδηγό ορθής διοικητικής πρακτικής θα έπρεπε να τον είχε εκδώσει η Κομισιόν. Ε, δεν το έκανε, ευτυχώς το έκανε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Είναι θετικό λοιπόν το ότι υπάρχει αυτός ο οδηγός και ελπίζω η Κομισιόν να φροντίσει να εκδώσει κάτι το νομικά δεσμευτικό και στον τομέα της διαφάνειας. Βεβαίως ε, δεν σημαίνει πως ε, χωρίς αυτό θα είχαμε λιγότερη ε, διαφάνεια. Για την επόμενη λοιπόν δεκαετία θα ήθελα η Κομισιόν να κάνει κάτι και να φροντίσει περισσότερο τον τομέα της διαφάνειας. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των Πρασίνων για δύο λεπτά η κυρία Άουκεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη για την εξαιρετική αυτή έκθεση και να τονίσω ότι υποστηρίζουμε τον διαμεσολαβητή και το έργο του γιατί καλό είναι να υπάρχει και ένας κανονισμός και όχι μόνο ένας οδηγός σε σχέση με τις υποσχέσεις προς τον πολίτη δύναμη των συνθήκων. Πρέπει να βελτιώσουμε παντού την κατάσταση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν κανονισμό και όχι έναν απλό οδηγό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί η έκθεση υποστηρίζει τα όσα ελέγχθησαν ως προς την παρουσία του διαμεσολαβητή και το έργο του. Θα πρέπει ο πολίτης να είναι στο επίκεντρο αυτής της υπηρεσίας δεν πρέπει να θεωρείται ο πολίτης ως εχθρός ε, έναντι του οποίου θα πρέπει να οχυρωθούμε. Γιατί η Επιτροπή πολλές φορές θεωρεί τον πολίτη ως ε, εχθρό. Έτσι τον αντιμετωπίζει. Ο κύριος Σεύκοβιτς μας είπε πολλά ωραία λόγια. Δεν αρκούν όμως. Χρειαζόμαστε πράξεις. Καλύτερα λοιπόν θα ήταν να είχαμε υπαλλήλους, να έχουμε υπαλλήλους της Επιτροπής που να σέβονται την εργασία τους και να καταπολεμήσουμε τη ε, διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός προς το πολίτη και διαφάνεια των κανονισμών. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι πολλές καταγγελίες προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες και όχι άλλες. Αυτό ανέφερε και η Επιτροπή Αναφορών. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πολύ δραστηριοί πολίτες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σωρία προβλημάτων. Πρόκειται για μια κοινωνία των πολιτών που θα πρέπει να υποστήριξουμε δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε γρήγορα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη, την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών για το έργο της. Νομίζω ότι διεξοδικά ασχολείται με τα θέματα που μας απασχόλησαν με βάση την ετήσια έκθεση και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Διαμαντούρο για την εξαιρετική συνεργασία. Όλοι θα πρέπει να επαυξήσουμε το ρόλο των πολιτών, γιατί όλες οι αναφορές σχετίζονται με αυτό το ε, παραγωγικό ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο δεν είναι πάντα αλληλέγγυο. Πολλοί ταπεινώνονται, δεν έχουν απασχόληση, κινούνται προς την φτώχεια. Γι' αυτό σε αυτή την περίοδο κρίσης θα πρέπει όλοι να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο διαφανής για να δίνει τάχιστα απαντήσεις προς τους πολίτες που διανύουν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαβράκος για δύο λεπτά κύριε πρόεδρε χαίρομαι ιδιαίτερα ότι εκπροσωπώντας την τελευταία πτέρυγα της βουλής διαπιστώνω πλήρη ομοφωνία στην αναγνώριση του έργου του κυρίου διαμαντούρου και στην εξαιρετική συνεργασία του με την επιτροπή αναφορών. έπαινοι ανήκουν στον κύριο διαμαντούρο που εκπροσωπεί και υπηρετεί επάξια ένα θεσμό συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με την έκθεση του Μεσολαβητού, καταχωρήσαν 2.510 αναφορές το 2011, ενώ ο θεσμός βοήθησε άμεσα περισσότερους από 22.000 πολίτες. Πολύ καλή η επίδοση αυτή. Πιστεύω όμως ότι πρέπει με κατάλληλο τρόπο ο θεσμός αυτός ο σημαντικός αυτός θεσμός να γίνει ευρύτερα ε, ε, γνωστός στους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση του ευρωβαρόμετρου το 42% των ευρωπαίων πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ένωσης. ο θεσμός είναι απαραίτητος και η άσκηση του θεσμού αυτού μέχρι σήμερα είναι επιτυχής όπως κάθε χρόνο βεβαίως οι περισσότερες έρευνες που διενεργήθηκαν από τον διαμεσολαβητή αφορούσαν την ευρωπαϊκή επιτροπή το 58 περίπου και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σχεδιαστούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με την επιτροπή προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της κρίσης των θεσμών και των δημοκρατικών αξιών συγχαίρω τον κύριο διαμαντούρο για τον εξαιρετικό τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του και συγχαίρω επίσης και την κυρία ματσόνη πρόεδρο της επιτροπής αναφορών που συνδράμει στην καλή συνεργασία των δύο οργάνων. με δε της ευκαιρίας να δώσω έναν τόνο αισιοδοξία και να πω ότι η κρίση θα περάσει. πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπέκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα κύριε Διαμεσολαβητή, αγαπητοί συνάδελφοι. Η, δραστηριότητα, η έκθεση δραστηριότητα κυρίας Ματσόνη αποδεικνύει πως πρέπει να ευχαριστήσουμε τον διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες του προς τον Ευρωπαίο πολίτη και για την πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά την Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα το οποίο παρακολούθησα. Στην Επιτροπή Αναφορών, ε, πέραν από τις 1.800 ε, ε, περίπου αναφορές, έχουμε μια ειδική έκθεση που αφορά τα παράπονα της καταγγελίες κατά της Κομισιόν και παρακολούθησα πως σε 16 χρόνια μόνο 18 φορές έγινε χρήση αυτού του συγκεκριμένου μέσου και παρακολούθησα πόσο επαγγελματικά διαχειρίστηκε ο διαμεσολαβητής ε, το θέμα αυτό με την ομάδα του. Παρά όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πτυχές ε, που παρατήρησα. Το ένα αφορά την ε, πληροφόρηση και επικοινωνία η οποία μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Εδώ πέρα θεωρώ πως το 27% των καταγγελιών που επεξεργάστηκαν που όντως ε, έγιναν δεκτές σημαίνει αντιστρόφως πως 3 τέταρτα δεν ε, απευθυνθήκαν σωστά και άρα πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη πληροφόρηση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάτι το οποίο υπάρχει στην Αυστριακή ε, δημόσια τηλεόραση και είναι μια εκπομπή σχετικής ε, πληροφόρησης. Το άλλο αφορά τον κανονισμό ε, για τον οποίο δημοσιεύσατε. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικά ελάχιστες προδιαγραφές για τη διοικητική πρακτική. Εδώ πέρα ξέρω πως δραστηριοποιείται ο κύριος Διαμεσολαβητής και του εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση του 2011 του διαμεσολαβητή σχετίζεται με πληροφορίες και βοήθεια κατά άμεσο τρόπο, καθώς και συνεργασία με τους εθνικούς συνηγόρους, έτσι ώστε να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα ως προς τους καταγγέλλοντες. Το 2011 ο διαμεσολαβητής βοήθησε περισσότερο από 22.000 πολίτες, μεταξύ των οποίων 2.510 υπέβαλαν καταγγελίες και 1.284 ζήτησαν πληροφορίες, καθώς και 18.274 ε, έλαβαν πληροφορίες διαμέσου του διαδραστικού οδηγού από την ιστοσελίδα του διαμεσολαβητή. Σε πάνω από 65.000, 65 ε, των καταγγελιών του 11 βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για τα δικαιώματα, την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των πολιτών και το γεγονός ότι το 61% έχει υποβληθεί, των ετοιμάτων ε, υποβλήθηκε μέσω ίντερνετ, δείχνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή χρήση του διαδικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Βαλέσα για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, το ποσοστό των καταγγελιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή ήταν αρκετά χαμηλό το 2011. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πιο γνωστό το θεσμικό αυτό όργανο στους πολίτες και βεβαίως να γίνουν πιο στενοί δεσμοί με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και με την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να συνεργάζεται ως το δυνατόν πιο στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα. Στηρίζω τον διαμεσολαβητή υπό την έννοια ότι η καλή διοίκηση δεν περιορίζεται μόνο στις νομοθετικές διατάξεις τα θεσμικά όργανα δεν πρέπει απλώς να σέβονται τις, νομ... υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νόμο, αλλά θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσία στους πολίτες, ώστε όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται σωστά και να χαίρουν σωστά, τον... να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους. Για ένα λεπτό, κυρία Πρέβεγκάστ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ευπρόσδεκτη η έκθεση των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Παραδέχομαι ότι ο θεσμός αυτός έχει σημαντικό ρόλο στην, στην βελτίωση των, της υπηρεσίας αλλά ε, πρόσφατα είχαμε το θέμα του Επιτρόπου Ντάλι και την περασμένη εβδομάδα, όσον αφορά τις προτάσεις για την ε, βελτίωση της Όλαφ, αναφέρθηκαν ε, τα διαδικαστικά δικαιώματα του ε, καταστατικού χάρτη. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν σκοπεύει να μελετήσει τις προϋποθέσεις ο διαμεσολαβητής γύρω από τις έκθεση, έκθεση της Όλαφ για την οδηγία ΤΑΚΟ όσον αφορά την ακαιρεότητα της διαδικασίας αυτής. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ματσόνη για την εξαιρετική και τη λεπτομεριακή αυτή εργασία καθώς και τον κύριο Διαμαντούρο για τη δραστηριότητά του κατά το έτος 2011. Έπεσε ο αριθμός των καταγγελιών και ο διαμεσολαβητής κατάφερε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με την κακοδιαχείριση θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ε, καταγγελιών που δεν ε, άπτεται της αρμοδιότητας του διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να δούμε πώς οι καταγγέλλοντες μπορούν να στραφούν προς το σωστό φορέα εκεί που δεν υπάρχει αρμοδιότητα του διαμεσολαβητού. Χαίρομαι διότι η υπάρχει μεγάλη και υψηλή συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητή και εθνικών συνηγόρων του πολίτη. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν για μία ακόμα φορά θέλω να αναφερθώ στην καλή συνεργασία που είχαμε με τον Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών γιατί επιδιώκουμε όλοι μαζί ένα πολύ σημαντικό στόχο να προσφέρουμε μια πραγματικά καλή δημόσια υπηρεσία εκ μέρους της Ευρώπης προς τους πολίτες. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε ότι ο αριθμό των καταγγελιών μειώνεται. Επίσης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για μας η καλή διοικητική συμπεριφορά, η δημόσια διοίκηση και ο σεβασμός τη είναι μια σημαντική αρχή που και την εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας δουλειά. Ακούστηκαν πολλά σχετικά με τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι πάντοτε μπορούμε να βελτιωθούμε. Και σαφώς και φέτος μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είμαι όμως πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία από τις ε, διαφανέστερες δημόσιες διοικήσεις της Ευρώπης και του κόσμου. Το πώς πρόκειται να βελτιωθούμε, πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας. Θα συνεχίσουμε με εντατική εσωτερική κατάρτιση των στελεχών μας θα αυξάνουμε συνεχώς την ευαισθητοποίηση για τις αρχές της καλής διοικητικής συμπεριφοράς και της διαφάνειας. Αυξάνουμε τη χρήση άτυπων διαδικασιών που πολύ συχνά μας βοηθούν να καταλήξουμε σε φιλικούς διακανονισμούς χωρίς ε, το περιττό γραφειοκρατικό βάρος. Επιδιώκουμε περισσότερους φιλικούς διακανονισμούς και σε αυτό μας συμβουλεύει πολύ καλά και ο ίδιος ο διαμεσολαβητής. Έτσι λοιπόν η καλή συνεργασία με εσά και το, τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε σε αυτό το τομέα της διαφάνειας. Θεωρώ ότι και εδώ τα τελευταία δύο χρόνια ε, καταβλήθηκαν σοβαρές προσπάθειες και από κοινού πετύχαμε πολλά. Ας πούμε, το κοινό μητρό διαφάνειας. Σπάνια υπάρχει τέτοιο στις πρωτεύουσε ε, των χωρών όλου του κόσμου. Κάτι παρόμοιο υπάρχει στη Ουάσιγκτον, ίσως και στη Βιέννη. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτό το μητρό λειτουργεί και όλο και περισσότερες ε, επιχειρήσεις θέλουν να εγγραφούν. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστώ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών για να αυξηθεί η συμμετοχή ε, της ε, ε, ε, του θέματος με τις δικηγορικές εταιρείες να δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα στην έκθεσή μας και πώς θα λειτουργεί αυτό το μητρό διαφάνειας. Είμαστε πιο διαφανείς από ό,τι παλαιότερα όταν ας πούμε στην περίπτωση της, ε, των, των μητρών επιτροπολογίας για το πώς συντάσσονται ποια είναι τα θέματα και το αποτέλεσμα των συζητήσεων, τα πρακτικά των συζητήσεων και όλα αυτά νομίζω ότι προχωρούν και μας βάζουν σε πολύ καλή θέση σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Τώρα, Έχουμε τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Δείχνουν ότι η διαφάνεια είναι σημαντική και πολύ συχνά οι Ευρωπαίοι πολίτε απογοητεύονται. Πρέπει όμω να αισθανόμαστε και περήφανοι και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είμαστε τα θεσμικά όργανα που περισσότερο εμπιστεύονται οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το συγκρίνουμε αυτό παρά την κρίση, το πόσοι οι πολίτε εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό είναι αρκετά ψηλότερο από ότι η εμπιστοσύνη προς τα εθνικά τους θεσμικά όργανα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Όσον αφορά την κατάσταση την περίπτωση του κυρίου Ντάλη και είμαι σίγουρος ότι και ο διαμεσολαβητής θα απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Θέλω να σα διαβεβαιώσω όλους ότι και στα ευρήματα της Όλαφ ήταν απόλυτα σαφές ότι η υπηρεσία είναι καθαρή σύμφωνα με την Όλαφ. Δεν υπήρχε περιστατικό που να αφορά την καλή λειτουργία και, την αποτελεσματική, ε, ε, και τον αποτελεσματικό χειρισμό των θεμάτων από τη Γενική Διεύθυνση και αυτό ε, αφορά επίσης και την οδηγία για τον καπνό. Και επίσης η οδηγία του καπνού θα, τεθεί, θα δοθεί ως πρόταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Είναι θέμα δύο-τριών εβδομάδων και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η οδηγία για τον καπνό θα ε, συζητηθεί, θα ψηφιστεί από αυτό το σώμα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και αφού σας υποβάλουμε την πρόταση όλοι θα συμφωνήσετε ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξη γιατί αυτό είναι σημαντικό θέμα για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους κυρίους και τις κυρίες βουλευτές που έλαβαν το λόγο και μίλησαν με καλά λόγια. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την στήριξή σας και γνωρίζουμε το ότι η δική σας στήριξη και η καλή σας δουλειά αυξάνει την ευθύνη που φέρουμε στους ώμους μας για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Αναφορών για να εξυπηρετούμε τους πολιτές ακόμα καλύτερα. Οπότε σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και την ενθάρρυνση να πω πως κάποιοι ευρωβουλευτές έθεσαν το θέμα του χαμηλού αριθμού καταγγελιών, μάλλον του χαμηλού, του υψηλού αριθμού καταγγελιών που δεν έγιναν δεκτές κ. Βαλένση νομίζω μεταξύ άλλων. Κοιτάξτε, πρέπει να τονίσουμε πως ε, λόγω του διαδραστικού οδηγού που έχουμε εδώ και τρία χρόνια στην ιστοσελίδα μας έχουμε το εξή καλό αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έρχονται σε εμά μόνο για του σωστού λόγου και όχι για λάθο λόγο. Το κοινοβούλιο αυτό εδώ και χρόνια επέμενε πως θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των μη αποδεκτών καταγγελιών. Το κάναμε αυτό σε σημαντικό βαθμό και Μάλιστα είμαστε ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για το ότι πρότεινε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Μποστινάρου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια και τη στήριξή σας. Να πω επίσης, γιατί ξέρετε, πως υπάρχει μια επαγγελματική διαστροφή του διαμεσολαβητή και προσπαθεί να είναι δίκαιος. Και για να είμαι δίκαιος πρέπει να πω πως πράγματι η Κομισιόν έχει τον υψηλότερο αριθμό καταγγελιών, όπως είπε και ο Επιτροπός είναι 65% ε, ούτως ή άλλως των υπαλλήλων της Ένωσης, αλλά εάν δείτε τις υποδειγματικές περιπτώσεις, τις 10 υποδειγματικές περιπτώσεις που βγάλαμε πέρσι, 5 υποδειγματικές περιπτώσεις για πραγματικά υποδειγματική επίδοση αφορούσαν την Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν τα προβλήματα συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν για τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως προσπαθούν και κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Κυρία Άουκεν, σας είμαι ευγνώμων, γνωρίζετε την άποψή μου για το θέμα του κανονισμού. Ήμουν και στο σπίτι το δικό σας και στο σπίτι της κυρίας Γιατερμάκη και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Άσταλα από την υπηρεσία ε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Να πω επίσης ε, στην κυρία Γκράστ να σας συγχαρώ για την απόφαση του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου χτες για την ε, σημαντική επέκταση των αρμοδιοτήτων ε, του, της ε, Ιρλανδής Θεμεσολαβητού καθώς 149 ε, φορείς υπήρχαν σε αυτήν και θα ήθελα μέσω ημών να μεταφέρω την ικανοποίησή μας. Όσον αφορά το ερώτημά σας, κυρία Πρέντεργαστ, για την οδηγία, η απάντηση είναι πως ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καταγγελία για την οδηγία αυτή. Εάν λάβουμε κάτι, βεβαίω θα πρέπει να φροντίσουμε πως πριν απευθυνθεί κάποιος σε εμάς, κάποιος καταγγέλων, θα είχε απευθυνθεί στον Όλαφ. Έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την εμπλοκή οποιοδήποτε θεσμικού οργάνωση στην περίπτωση αυτή της Κομισιόν δηλαδή. Τέλος, θα ήθελα και πάλι να αναγνωρίσω την προσφορά του Επιτρόπου του κ. Σεύκοβιτς για την ορθή διοίκηση. Το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και βεβαίω ε, αναμένουμε τη στενή μας συνεργασία και βεβαίω σημειώνουμε την αύξηση της συνεργασίας της Κομισιόν για να βρίσκουμε φιλικές λύσεις μέσω άτυπων διαδικασιών, κατά το οποίο είναι καλό για εσάς, για εμάς και πάνω απ' όλα για τους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διαμαντούρο. Η κυρία Ματσόνη. Ε, εκτίμησα ιδιαίτερα την απόψινή συζήτηση. Νομίζω ότι αποδεικνύει άμεσα ε, για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν πολύ καλά δίκτυα συνεργασίας ε, της κοινωνίας των πολιτών και αγαστή συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και άλλων φορέων καθώς και του διαμεσολαβητή και επίσης πώς όλοι συμμεριζόμαστε του στόχους αυτής της επίπονης εργασίας. Πρόκειται για μία όσμωση μεταξύ των δύο οργανισμών που μας βοηθούν θα αναλάβουμε λάβουμε υπόψη τις καλύτερες εμπειρίες των μεν από τους δε και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα να παρεμβαίνουμε μέσω των νέων μέσων τεχνολογίας. Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει υπόψη και τις ε, σχέσεις μας σχέσεις παρακολούθησης των ε, πολιτών ενώ πολλές φορές ε, απευθύνονται στο διαμεσολαβητή. E ενώ πολλές φορές ε, λαμβάνουμε υπόψη ότι οι πολίτες απευθύνονται στο διαμεσολαβητή, ενώ θα έπρεπε να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών. και πολλές φορές οι καταγγελίες μπορούν να πλήξουν τον οποιονδήποτε. Μία καταγγελία μάλιστα ε, έπλητε τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σεύκοβιτς και είμαι πεπισμένη ότι οι στόχοι αυτοί είναι ευκταίοι από κάθε πλευρά. Παρά τις καλές μας προθέσεις βεβαίως δεν υπάρχει επαρκής ρυθμός σπουδής από Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχει απλούστευση και άμεση αντίδραση όπως θα επιθυμούσαμε και αυτό το βλέπουμε και στα δικά μας αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών αλλά και στις καταγγελίες που λαμβάνει ο διαμεσολαβητής. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Σεύκοβιτς ενδιαφέρεται βεβαίως και θα προωθήσει το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύριο θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή στις 11.30. Τώρα διακόπτουμε τη σύνοδο η οποία θα επαναληφθεί στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστώ.